Έκλεισε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Αύριο το πρωί θα γίνει η επόμενη α, συνεδρίαση από τις 10 έως τις